Start. Να ξεκινήσουμε. We should, uh, take your seat. Καθίστε παρακαλώ. Φροντίστε να έχετε τις κάρτες σας, τις μηχανές. Δεν θα ελέγξουμε βασιζόμαστε στον επαγγελματισμό των τεχνικών μας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα ψηφίσουμε για τον δημοσιονομικό έλεγχο της βοήθειας στο Αφγανιστάν, έκθεση για την ΜΑΚΙ. Οπότε, τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 6. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Πρέπει να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Ωραία, πέρας. Δεκτή. Οχτώ. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9. Αφγανιστάν. Το Αφγανιστάν ψηφίζουμε. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 12 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 κατά απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21, 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μπορούμε να την επαληθεύσουμε αν θέλετε. Απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία η ηλεκτρονική άρτη ψηφοφορία πέρας Ωραία. 32 υπέρ. Τέσσερις αποχές. Συγχαρητήρια στην κυρία Γιάννη Μάκη. Λοιπόν, Γεωργία. Έκθεση Λίζεκ. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Εντάξει, να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 με προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 23. Και πέρασε. Απορρίπτεται με μια ψήφο διαφορά. Κινητοποιηθήκατε, αλλά περνάμε στην επόμενη. Η 24-25. Υπέρ κατά αποχές δεκτή η 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 29 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε. Την 29 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Μάλιστα δεκτή. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Μάλιστα, να επαληθεύσουμε την 30. Άρχεται την ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Αυτό είχα δει και εγώ από εδώ πάνω. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 32 υπέρ. Κατά αποχές να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 32. Και πέρασε. Απορρίπτεται λοιπόν. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 38 υπέρ. Κατά. Α... Αποχές. Να υπαλληθεύσουμε. Την 38 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή λοιπόν με τέσσερις ψήφους φορά Να ξανά επαληθεύσουμε. Λοιπόν, 39 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω πως απορρίπτεται να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 40. Πέρας. Δεκτή. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε και πάλι. 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή με δύο ψήφους διαφορά. 42 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε. 42. Άρχεται η ψηφοφορία. So, vote is... Πέρας. Απορρίπτεται με ισοψηφία. Σαράντα τρία υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή νομίζω. Να επαληθεύσουμε. 43. Νομίζω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πέρασε. Δεκτή. Περνάμε στην 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 45 υπέρ. Κατά. Νομίζω πως έγινε δεκτή. Να υπαλληθεύσουμε την 45 άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Όχι. Α, με την ψήφο του κυρίου Σβόμποντα γίνεται δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 47 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Να την επαληθεύσουμε. Ωραία. 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή λοιπόν. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 49 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 53 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως πρέπει να επαληθεύσουμε την 53 άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 54 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 58 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω πως πρέπει να την επαληθεύσουμε. 58 Άρχεται η ψηφοφορία. Έρας. Δεκτή. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Εκτιμώντας α. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ε, υπαριθμόν 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε. Άρχεται ψηφοφορία για την 2. Πέρας. δεκτή και με τη δική σας ψήφο. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, δεκτή. 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7 και 8 σε δύο μέρη. Α, όχι μαζί. Ωραία. Ταυτόσημες. Υπέρ κατά αποχές δεκτή παριθμών 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές Νομίζω πως έχει απορριφθεί να την επαληθεύσουμε. 12. Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Συν 2 ψήφι κατά. Γίνεται δεκτή λοιπόν. Περνάμε στην Θέλετε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Α, από 1 μέχρι 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. Η 8 καταπίπτει, οπότε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Α, παράγραφος 8. Λοιπόν, ψηφίζουμε... Μα αυτή εάν δεν έχει υιοθετηθεί η συμβιβαστική 5. Γι' αυτό, γιατί η 5 είχε γίνει δεκτή, οπότε προσπεράσαμε την 8. Ο συνήθως είχαμε δίκιο. Λοιπόν, τώρα άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υπάρχουν δύο άτομα ακόμα που πρέπει λοιπόν να ψηφίσουν. Χάνε Βόμποντα και κάποιος άλλος ήταν εκεί. Πέρας, ωραιότατα, εγκρίθηκε συγχαρητήρια στον κύριο Λίζακ. Okay. Yeah. Now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 την αίτηση της Κροατίας για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, όσοι θέλουν να φύγουν ήρεμα και οι υπόλοιποι ας μείνουν. Έχουμε λοιπόν την συνθήκη για την ένταξη της Δημοκρατίας της Κροατίας ας λάβουμε υπόψη πως για την Κροατία και για την Ένωση είναι μια σημαντική στιγμή και ας συμπεριφερθούμε αναλόγως. Τα δε σημεία 7 και 8 θα συζητηθούν μαζί καθώς έχουμε συνθήκη προσχώρησης και την ίδια την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας και οι δύο αφορούν την Κροατία και οι δύο είναι εκθέσεις του κυρίου Σφόποντα. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν διαπραγματεύσεις 30 Ιουνίου. Το Συμβούλιο ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την συγκατάθεσή του. Η υπογραφή της συνθήκης έχει προγραμματιστεί για τις 19 Δεκεμβρίου στη Βαρσοβία και μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία κύρωσης στα κράτη-μέλη και την Κροατία με στόχο να ενταχθεί 1η Ιουλίου 2013 το 28ο κράτος μέλος. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε την συγκατάθεσή μας. Τώρα θα ζητήσω από τον κύριο Σοβοντάν να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, μιλάμε για τα σημεία 7 και 8. Ο σημείο 8 είναι, αν θέλετε, το σοβαρότερο, αλλά και το απλούστερο είναι για ένα ναι ή όχι. Η σύστασή μου είναι βεβαίως ναι για την προσχώρηση της δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θυμάστε πως ήταν μακροσκελής Η διαπραγματεύσεις πάντα σας ενημερώναμε και παρακολουθούσαμε και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια τις διαπραγματεύσεις. Είπαμε που πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις. Το κοινοβούλιο μας τήρησε μια στάση η οποία παρακολουθούσε πάντα θετικά αλλά και με κριτική ματιά τη διαδικασία για να ενθαρρύνουμε την διαδικασία στην ένταξή της. Εμείς ως κοινοβουλία. καταλήξαμε στο ότι αντί για το 2009, το 2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία και θα μπορέσουμε εντός αυτή τη θητείας του Κοινοβουλίου, δηλαδή το 2013, να ενταχθεί αυτή η χώρα. Και άρα μπορούμε να λάβουμε αυτή την απόφαση, δηλαδή να συμφωνήσουμε στη σύμβαση έτσι ώστε, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος της 19 του μηνός να υπογραφεί η ε, ένταξη στην ε, Βαρσοβία. Βεβαίως ε, τα ουσιαστικά έχουν εκπληρωθεί ώστε θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Εγώ πάντα τόνιζα πως το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την Κροατία αλλά ολόκληρη την περιοχή αν και ξέρουμε πως η επόμενη ένταξη ε, θα πάρει χρόνια γιατί βεβαίως ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με κάποια χώρα της περιοχής. Θα δούμε τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο αλλά υποθέτοντας πως ε, θα διαπραγμα... θα... οι διαπραγματεύσεις θα διαρκέσουν τόσο πολύ όσο με την Κροατία τότε τα επόμενα λίγα χρόνια δεν θα έχουμε κάποια ένταξη από αυτή την περιοχή αλλά βεβαίως αυτό σημαίνει και γι' αυτό είναι το σημαντική απόφασή μας πως δεν είναι αυτό το τέλος της διαδικασίας, αλλά πως δίνουμε ένα πράσινο φως για την ένταξη αυτής της περιοχής, αλλά και αυτό μας διδάσκει η περίπτωση της Κροατίας, πως η κάθε χώρα πρέπει να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις στο εσωτερικό της για να υπάρξει ένταξη. Οπότε η σύστασή μου είναι ναι στην ένταξη και νομίζω πως έτσι θα δώσουμε την σωστή κατεύθυνση που πρέπει. Όμως θα ήθελα ταυτόχρονα να προτείνω στο Κοινοβούλιο να έχουμε ένα συνοδευτικό ψήφισμα στο οποίο θα αναφέρουμε το τι πρέπει ακόμα να κάνει η Κροατία. Δεν βλέπω καμιά ιδιαίτερη δυσκολία βεβαίως στη διαδικασία κύρωσης, αλλά αυτό προϋποθέτει πως η Κροατία θα κάνει τα απαραίτητα βήματα μεταρρυθμίσεων στον τομέα της δικαιοσύνης, ε, στην οικονομική και κοινωνική πολιτική και πως η Κροατία όσον αφορά τα πολιτικά δικαιώματα και τα αστικά δικαιώματα τα δικαιώματα των μειονοτήτων ε, και δεν μιλάμε μόνο για τη σερβική μειονότητα αλλά μειονότητες όσον αφορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό, οτιδήποτε ε, είναι μειοψηφία στην κοινωνία γιατί γνωρίζουμε πως υπήρχαν κάποια περιστατικά που δεν είναι θετικά και στα οποία ασκήσαμε κριτική. Υποθέτω λοιπόν πως θα ε, κάνει τα απαραίτητα η Κροατία για να αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα. Έχουμε λοιπόν αυτό το ψήφισμα και θα καταθέσουν και κάποιες άλλες επιτροπές τροπολογίες που θα ξεκαθαρίσει πως ναι, πρέπει να γίνει η ένταξη, θέλουμε μια γρήγορη διαδικασία κύρωσης, αλλά και η Κροατία θα πρέπει να έχει κατά νου την ευθύνη της για ε, συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, μέχρι επιστροφή των προσφύγων, μέχρι ζητήματα εσωτερικής αγοράς, μέχρι ακόμα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, ε, μέχρι άλλα ζητήματα. Όπως είπα, πολιτική διακρίσεων πρέπει να κάνει κάποια βήματα η Κροατία. Όχι μόνο η Κροατία. Γνωρίζουμε πως σε κάποια κράτη-μέλη έχουμε προβλήματα, αλλά η Κροατία είναι τώρα στη διαδικασία της ένταξης και πρέπει να φροντίσει αυτά τα πράγματα. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, υποβάλλω προς συζήτηση την έκθεσή μου Ελπίζω να μπορέσουμε να εργαστούμε τόσο γρήγορα ώστε στις 20 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο στην Επιτροπή να ψηφίσουμε και μετά στην πρώτη Ολομέλεια του Δεκεμβρίου να λάβουμε και την ανάλογη απόφαση. να συμφωνήσει δηλαδή και το Κοινοβούλιο και θα ολοκληρωθεί έτσι μια διαδικασία η οποία διάρκησε πολύ αλλά ε, νομίζω πως ε, χαρακτηρίστηκε από αμοιβαία θετικά αισθήματα και σεβασμό και στην Κροατία πάντα ε, σέβονταν αυτά τα οποία έχει να πει το Κοινοβούλιο γιατί όπως είπα υπάρχουν αμοιβαία θετικά αισθήματα αλλά και η απαραίτητη κριτική και ελπίζω λοιπόν να αποτελέσει αυτό ένα θετικό παράδειγμα των σχέσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποψηφίου χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζετε νομίζω πως αυτό είναι ένα καλό σημάδι όχι μόνο για εμάς αλλά και για τις υποψήφιες χώρες στην περιοχή και γενικά γιατί Μπορούμε έτσι να δείξουμε πως τα πράγματα συνεχίζονται και δεν σταμάτησε η διαδικασία της διεύρυνσης και για την Κροατία. Αναμένουμε την ένταξη και τους συναδέλφους μας που θα γίνουν βουλευτές στο συντομότερο δυνατόν τώρα. Θα ζητήσω από τον κύριο Πόσελτ που είναι σκιώδης ηγητής να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να θέσω το ερώτημα πότε θα γίνει η ψηφοφορία ακριβώς στο Στρασβούργο, γιατί το είχαμε πει αρχικά για 14 στη Δευτέρα. 20 θα είναι Κυριακή. Α, Πέμπτη. Πέμπτη λέει ο κύριος Βόμποντα. Α, κοιτάξτε. Εντάξει, Παρασκευή και Σάββατο, αλλά να μείνουμε, αλλά το, η Κυριακή παραπάει. Αν και βεβαίως πρόκειται για τα 91 τα γενέθλια της γέννησης του ο το Φον Νομίζω θα ήταν και μια συμβολική ημερομηνία για την επανένταξη της ε, Κροατίας. Οπότε πέμπτη είναι 17 του μηνός, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι, βεβαίως. 17 του μηνός, συμβαίνει και ο κύριος Φόβοντα. Ε, να σοβαρευτούμε τώρα. Ως ε, πρεσβύτερος των σκιωδών εισηγητών, να ευχαριστήσω τον κύριο Σβόμποντα για την ε, πολυετή συνεργασία και πολύ καλή συνεργασία για την προετοιμασία της ένταξης της Κροατίας. Είναι πραγματικά ιστορική στιγμή, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε εύκολα τη λέξη ιστορικός, αλλά πριν από 20 χρόνια ε, ήμουν εγώ στην Κροατία, ο πόλεμος τότε ήταν κτηνόδης και πάνω από 100.000 άνθρωποι το φθινόπωρο του έτους 91 εκδιώχθηκαν, το Βούκοβαρ καταστράφηκε μία τότε πολύ ζωντανή ευρωπαϊκή πόλη και αν ζούσε κανείς τότε τους 10.000 νεκρούς, τους πάνω από 100.000 εκδιωγμένους και το να μπορέσει μετά από αυτό να βοηθήσει κανείς την ένταξη της Κροατίας είναι κάτι το οποίο τον κάνει να λέει τη λέξη ιστορικός. Και χαίρομαι για το ότι καταφέραμε να ενταχθεί η Κροατία. 20 χρόνια χρειάστηκε και θα ήθελα να πω πως χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι κατάφερε η Επιτροπή μας και καταφέραμε να πάει και στην Ολομόλια, το είπε και ο κύριος Σβόμποντα, μίλησε για το 2009, να α, καταφέρουμε κάποια πράγματα. Ήταν άνθρωποι που ήταν κατά. Και αν δεν ορίσαμε, αν δεν ορίζαμε και κάποιες ημερομηνίες, γιατί βεβαίως τα κριτήρια εκπληρώνονται και πρέπει να υπάρχουν και κάποιες ημερομηνίε και αν δεν ασκούμε πίεση δεν συμβαίνει τίποτα και αναβάλλονται τα πράγματα για του Αγίου ποτέ. Οπότε Οφείλεται αυτό βεβαίως κατά κύριο λόγο στους κοράτες τους ιδίους και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί υπήρχαν πάρα πολλά εμπόδια για αυτή την πορεία και θα ήθελα να πω πως κανένας άλλος υποψήφιος δεν έπρεπε να αντιμετωπίσει τόσους πολλούς δίκαιους και αδικαιολόγητους όρους όπως η Οκρατία. Δηλαδή Καμιά φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριφέρονταν σαν μητέρα η οποία μεγάλωσε 7 παιδιά και στο 8ο παιδί έβγαζε το άχτη της και έκανε όσα δεν έκανε στην ανατροφή των υπολείπων 7. Οπότε, Σβόμποντα, ελπίζω να μην σε ταλαιπωρεί εκεί πέρα ο Μπροκ. Εγώ λοιπόν θεωρώ πως θα πρέπει να δούμε και το έχουμε συζητήσει αυτό, πως το ψήφισμα γιατί εντάξει στο διατακτικό συμφωνούμε θα πούμε ξεκάθαρα ναι όσον αφορά λοιπόν το ψήφισμα το οποίο το συνοδεύει βεβαίως να αναφερθούμε επικριτικά σε κάποια σημεία αλλά δεν θα πρέπει τώρα να μπούμε και να συζητάμε με το τι θεωρεί κάθε ομάδα εδώ πέρα μέσα στο Κοινοβούλιο σωστό και επιθυμητό. Όχι μόνο γιατί θα γίνει μετά τα σχηνοτενέ το ψήφισμα, ενώ θα έπρεπε να είναι σύντομα, αλλά και γιατί βρισκόμαστε και συνεδριάζουμε σε μια δύσκολη στιγμή. Δύο μέρες πριν από τις κροατικές εκλογές. Δεν θέλουμε να παρέμβουμε στα εσωτερικά λοιπόν της Κροατίας. Και λίγες εβδομάδες πριν από ένα δύσκολο δημοψήφισμα επίσης στην Κροατία. Και δεν θα πρέπει να πατρονάρουμε την Κροατία με πατερναλιστικό ύφος. Οπότε πρέπει να περιοριστούμε στην ουσία και να μην μπούμε στην εσωτερική πολιτική στο ψήφισμα αυτό και ε, προσωπικά έχω επεξεργαστεί μια σειρά τροπολογίες για την ομάδα μας που προσπαθούν να κάνουν το κείμενο κάπως πιο σύντομο αντί να το μεγαλώσουν κι άλλο. Οπότε όλες μου οι τροπολογίες είναι προτάσεις για να γίνει πιο σύντομο το κείμενο και θα το συζητήσουμε στη δεύτερη ανάγνωση αλλά ως βασική γραμμή ε, θα, αυτό θα συνιστούσα και στις άλλες ομάδες και αυτό το οποίο θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Σφόμποντα δεν το κατέστησα τροπολογία γιατί νομίζω πως μπορεί να το κάνει καλύτερα ο ίδιος ο εισηγητής του. Σημείο 16 το τέλος είναι σημαντικό γιατί λέει ξεκάθαρα πως χαιρετίζουμε υποστηρίζουμε την υπογραφή της συνθήκης ένταξης και πριν έχουμε το σημείο που χαιρετίζουμε την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και μετά περνάμε σε διάφορα αλλά και λέμε πως υπάρχουν τα χύψη προβλήματα. Αλλά πρέπει να πούμε πως έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις. Δεν μπορούμε να απαιτήσουμε ε, από την Κροατία κάτι παραπάνω από αυτό που απαιτούμε από τα κράτη-μέλη από τις άλλες υποψήφιες χώρες. Γι' αυτό προτείνω το σημείο 16 και το σημείο 1 να ενισχυθούν κάπως, να πάνε όλα μαζί στην αρχή για να φανεί το ναι το οποίο προτείνουμε και το ναι που λέμε το τάσετε υπέρ να μπει στην αρχή του κειμένου και μετά να αναφέρουμε τα διάφορα σημεία τα οποία αναφέρονται. γιατί εντάξει και οι δικές μας τροπολογίες είναι αρκετές, αλλά είναι κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν το κείμενο πιο μεγάλο. Εμείς όπως είπα προσπαθούμε να το συμμαζέψουμε. Αυτά λοιπόν για την πρώτη συζήτηση και όπως είπα και πάλι ευχαριστώ πολύ όλες τις ομάδες για την καλή συνεργασία. Well, thank you very much. And, uh, Σας ευχαριστούμε. κ. Μπάγκελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα επαναλάβω και εγώ τις θερμές μου ευχές και την ικανοποίησή μας για την εξέλιξη του θέματος ως τώρα. Συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι η Κροατία αξίζει να προχωρήσει μετά από αυτή τη μακρά διαδικασία διαπραγματεύσεων. Και επίσης Νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι σε αυτή τη διαδικασία η Κροατία αξιοποίησε όλες τις ευκαιρίες που δόθηκαν. Κάτι που εντόπισε ήδη και ο εισηγητής. Ωστόσο, θεωρώ ότι όλη η συζήτηση η σημερινή θα πρέπει να ολοκληρωθεί βάσει των ε, προτύπων που συνήθως ισχύουν εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο δικό μας χαρακτηριστικό είναι ότι μεταξύ των βουλευτών υπάρχουν κάποιοι ένθερμοι υποστηρικτέ της Κροατίας ενώ οι υπόλοιποι είναι απλώς φίλοι τη χώρα. Όλοι λοιπόν θέλουμε να προσχωρήσει η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι επίσημες διαδικασίες με έναν τρόπο στο δυνατόν πιο διαφανή και αποτελεσματικό όσο το δυνατόν συντομότερα και τώρα δεν θα ήθελα να αναγυροδέω ζητήματα τα οποία θα σφραγιστούν με τη λήξη των διαπραγματεύσεων. Νομίζω όμως ότι δεν θα ήταν κακό να σταθούμε σε ορισμένα σημεία. Σημεία τα οποία θα έπρεπε να λάβει υπόψη ένα νέο κράτο μέλο προκειμένου να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συγκεκριμένη περίσταση πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Κροατία πλήρωσε το τίμημα της προσχώρησης. Νομίζω λοιπόν δίκαιο είναι να έρθει όλη η διαδικασία σε αίσιο πέρα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μπρόκ τώρα. Κύριε Έλμαρ Μπρόκ. You have the floor, sir. He was speaking, you know, to friends. Ε, μιλούσα σε φίλους του στην Κροατία. Όχι, όχι, λέει ο κύριος Μπρόκ. Όχι, ήταν ε, βουλευτής από τη Γερμανία για τα οικονομικά. Ναι, ναι, όχι, κομματικός φίλος, όχι φίλος. Μία σύντομη παρατήρηση θέλω μόνο να κάνω. Πως πρώτον υποστηρίζω την έκθεση Σβόμποντα, δεύτερον στους σταθείς αυτούς καιρούς πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα και να πούμε ναι και πράγματι αναφέρεται πως πρέπει να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις σε κάποιους τομείς, ζητήματα διοίκησης, κράτους δικαίου, διαφθοράς, ε, εκεί που δεν είναι τα πράγματα ακόμα τελείως εντάξει, αλλά θεωρώ πως με, τα, με με αυτά τα οποία αναφέρθηκαν στην ενδιάμεση έκθεση της ε, Κομισιόν ε, στις 11 ε, Μαρτίου. Νομίζω πως έχουμε τις, να απαραίτητη εμπειρία για να προχωρήσουμε στην πορεία αυτή και νομίζω πως θα δούμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα κράτη της Βαλκανικής όπου θα έχουμε πάρα πολλά εμπόδια Ε, των Βαλκανίων που έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Μην ξεχνάμε πω η υπόσχεση ένταξη είχε δοθεί στην ε, Θεσσαλονίκη αρκετά παλιά και θα πρέπει νομίζω να δείξουμε πω ε, με την ένταξη της παραμένει η πόρτα ανοιχτή για τι βαλκανικέ χώρε για να υπάρξει μια σταθεροποίηση στην περιοχή και άρα νομίζω πω πρέπει να ακολουθήσουμε τη σύσταση του εισηγητή για να στείλουμε το σωστό μήνυμα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Now... Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος Κομισιόν, ο κύριος Λάγκερ, παρακαλώ, να λέει το λόγο. Äh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές. Όπως ξέρετε, η Κομισιόν ε, στις 12 Οκτωβρίου έδωσε την σύστασή της. Ήταν θετική και ο Επίτροπος Φίλε ήταν ε, στο Κοινοβούλιο στις 12 Οκτωβρίου για να την παρουσιάσει στο πλαίσιο του πακέτου διεύρυνσης. Όπως αναφέρθηκε ήδη η Κροατία είναι η πρώτη χώρα η οποία πέρασε τη νέα διαδικασία ένταξης και έπρεπε να εκπληρώσει πάρα πολλά πράγματα και κάποιοι είπαν πως διοίκησε λίγο περισσότερο αλλά βοήθησε για να οδηγηθεί η Κροατία στην οδό αυτή της ένταξης και η Κομισιόν ήταν πάρα πολύ θετική στην τελευταία της έκθεση αξιολόγηση και είπαμε πως είναι έτοιμη για να γίνει μέλος η Κροατία. Η έκθεση αυτή η προόδου θα είναι λοιπόν η τελευταία και τώρα θα συνεχίσουμε με κάποιες εκθέσεις, παρακολου... εκθέσεις παρακολούθησης. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για αυτές τις εκθέσεις παρακολούθησης γιατί η Κομισιόν έλαβε μια ισχυρή εντολή για την περαιτέρω προετοιμασία της ε, Κροατίας ε, για την ένταξη. Οπότε, όπως είπα, δεν θα υπάρξει νέα έκθεση προόδου. Θα έχουμε μια έκθεση παρακολούθησης, όπως λέγεται, το επόμενο φθινόπωρο που θα είναι κάπως διαφορετική θα μπαίνει δηλαδή περισσότερο σε λεπτομέρειες για τις υποχρεώσεις της Κροατίας και το ποια πρόοδος έχει σημειωθεί. Ως μέσο προετοιμασίας αυτής της έκθεσης χρησιμοποιούμε τους λεγόμενους πίνακες παρακολούθησης που τους επεξεργαζόμαστε κάθε εξάμεινο. Οι πίνακες αυτοί προετοιμάζονται μεταξύ άλλων με βάση πληροφορίες που λαμβάνουμε από την Κροατία αλλά και από μη κυβερνητικές οργανώσεις και από άλλους για να έχουμε μια δίκαιη αντικειμενική αξιολόγηση της προς ε, Κροατίας. Τους επόμενους λοιπόν πίνακες αυτούς θα τους υποβάλουμε τον επόμενο μήνα στο Συμβούλιο μαζί με την ε, έκθεση αυτή η Επίσης θα συνεχιστεί ο διάλογος που έχουμε με την Κροατία στη διαδικασία της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Υπάρχει και μια συνεδρίαση για τη συμφωνία αυτή το Δεκέμβριο. Ε, επιπροσθέτως, πέρα δηλαδή από αυτή την έκθεση και τους πίνακες που ανέφερα θα έχουμε εξαμηνιές εκθέσεις για τα κεφάλαια εκείνα τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα το περίφημο κεφάλαιο 23 περί δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλά και το κεφάλαιο του ανταγωνισμού και το κεφάλαιο 24 δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια επίσης Ε, η σύμβαση αναφέρει πως ε, το Συμβούλιο μπορεί να, να λάβει περαιτέρω μέτρα εάν δεν τηρηθούν όλες οι υποχρεώσεις της ε, Κροατίας και επίσης υπάρχει η δυνατότητα να αποστείλουμε τις λεγόμενες προειδοποιητικές επιστολές στην Κροατία εάν υπάρξουν προβλήματα στην έκθεση παρακολούθησης να ολοκληρώσω λέγοντας πως ο μηχανισμός αυτός ε, για μας είναι μια δυνατότητα να δούμε και να υπάρχει μια επαφή με τους Κροάτες για το πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω στην προετοιμασία και ο κοινό μας στόχος βεβαίως είναι η Κροατία να προετοιμαστεί πλήρως για να είναι έτοιμη όταν θα ενταχθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριο Σβόμποντα. Ευχαριστώ. Σύντομα θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και την Κομισιόν και το Συμβούλιο και τις διάφορες προεδρίες για το ότι συνεισέφεραν ε, με τη συνεργασία τους ε, με τη συνεργασία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κομισιόν όλα αυτά οδήγησαν λοιπόν στο να καταλήξουμε σε μια καλή λύση τώρα θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις η πρώτη αναφέρεται σε αυτό το οποίο προτείνει ο κύριος Πόσελτ για την ε, πρότασή του το άρθρο 16 και το άρθρο 1 να συγχωνευτούν, ε, δηλαδή τα κατά βάση θετικά άρθρα που λένε ναι και τα υπόλοιπα να γίνουν ένα άρθρο 2 έτσι ώστε και σε αυτή την έκθεση να είναι σαφές πως υποστηρίζουμε την ένταξη πως θα παρακολουθούμε βεβαίως ε, και μετά θα δούμε τι θα γίνει με τις τροπολογίες του κυρίου Πόσελτ περί συντόμευσης του κειμένου. Θα το δούμε αυτό με τους σκιώδεις εισηγητές. Θα καθίσουμε μαζί και θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιους συμβιβασμούς, συμβαστικές λύσεις. Και μετά να παρακαλέσω και τους συναδέλφους βεβαίως να στηρίξουν την έκθεση. Νομίζω πως θα είναι αυτό ένα σημαντικό μήνυμα. Επίσης, συμφωνήσαμε να δούμε τις εκθέσεις ε, παρακολούθησης και τις εξεμηνιαίες εκθέσεις, αλλά Όπως αναφέρθηκε ήδη, έβλε, εάν υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στις διαδικασίες της ε, μεταρρυθμιστικές, ε, νομίζω υπάρχει και η ομάδα εργασίας ε, Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά δεν θέλουμε τώρα μια μόνιμη παρακολούθηση από πλευράς Κοινοβουλίου. Αυτή είναι δουλειά της Κομισιόν. Μόνο εκεί όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Οπότε ευχαριστούμε. Και πάλι ευχαριστώ και πάλι τους και του συναδέλφους και ελπίζω βεβαίως ε, να υπάρξει συνένεση για να συμφωνήσουμε και στην έκθεση και στην συνθήκη. Και ε, συγγνώμη που ήθελα να κουβαλήσω τον κύριο Πόσελτ Κυριακή στο Στρασβούργο. Τε, ξέρω πως του αρέσει, αλλά τελικά θα ψηφίσουμε πέμπτη. Ευχαριστώ. Πριν ε, ολοκληρώσουμε, να σας ανακοινώσω πως η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι αύριο Παρασκευή 21 Οκτωβρίου μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Δεύτερη ανακοίνωση είναι πως ε, αποφασίσαμε να επεκταθεί η προθεσμία καταθέσεων τροπολογιών ε, για την Ουκρανία μέχρι την 5η 3 Νοεμβρίου το μεσημέρι. Οπότε κύριε Μπροκ, κύριε Πρόεδρε, μήπως γίνεται να το κάνουμε μέχρι τη Δευτέρα, τις 31 Οκτωβρίου. Μα εγώ είπα μέχρι το Νοέμβριο, 3 Νοεμβρίου. Α, 3 Νοεμβρίου. Α, μάλιστα. Ωραιότατα. Finally, we got agreement on this one. The third announcement is... Συμφωνήσαμε, ωραία. Επόμενη συνεδρίαση στο Στρασβούργο 24 από τις 7 και 4 μέχρι τις 9 και 4 παρουσία του Γάλλου Υπουργού Αμήνης και τελευταία ανακοίνωση να ανακοινώσω πως ε, ήταν η ικανοποίησή μου που προέδρευσα σε αυτή την ιστορική συνεδρίαση και να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και καλή επιτυχία στην Κροατία. Κύριε Σφόμποντα. Δεν ξέρω εάν ε, γνωρίζετε αν ο κύριος Μπρόκ θα παραμείνει στα αριστερά ε, στο μέλλον ή αν θα μετακινηθεί ξανά στο κέντρο. Νομίζω καλή ιδέα θα ήταν. Θα ενισχύσει και, το, και την αριστερά και το ΕΛΚ. Μα εάν είστε δεξιά μετά το μόνο επόμενο βήμα είναι στα άκρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε στο Στρασβούργο και συγχαρητήρια στους Κροάτες φίλους μας.